Θα σταματήσουμε για πολύ λίγο για να έρθει η Επίτροπος. Με την ησυχία σας, κύριε Επίτροπε. μη βιάζεστε. Okay, I think everyone is in place. Όλοι έφτασαν. Το επόμενο σημείο είναι μια η έκθεση της κυρίας Γκρέσλε για τη γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Όλαφ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε για τέσσερα λεπτά που είναι η συγκητριά μας. Κυρία Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή η μικρή αναθεώρηση της ε, οδηγίας της Όλαφ με την οποία ασχολόμαστε σήμερα το βράδυ ε, καταδεικνύει ότι είναι σε θέση να δράσουν σωστά και γρήγορα τα θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες. 12 εβδομάδες χρειάστηκε μέχρι να ε, γίνει η πλήρη επεξεργασία της έκθεσης. Και σας παρακαλώ λοιπόν αύριο να εγκρίνετε και ευχαριστώ λοιπόν την Επιτροπή και το Συμβούλιο και την Ολλανδική Προεδρία. Πραγματικά πάρα πολύ καλή επίδοση και πρέπει να την μιμηθεί σε άλλες περιστάσεις αυτή το Συμβούλιο η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει μια σημαντική αλλαγή, η οποία ε, είναι η εξή. Η Επιτροπή Αποπτίας της ΟΛΑΦ, η οποία ως τώρα ήταν ε, μέρος της ΟΛΑΦ, πλέον ε, αποδεσμεύεται και εντάσσεται στο οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ως τώρα οι υπάλληλοι αυτοί, τα πέντε αυτά υψηλόβαθμα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας ήταν ε, υποκείμενα. Προϊστάμενος τους ήταν ε, ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ, ακριβώς αυτός τον οποίο υποτίθεται θα έλεγχαν. Αυτή λοιπόν, αυτός ο κίνδυνος για τη σύγκρουση συμφερόντων και ε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι δυσνόητο και έτσι λοιπόν αυτό ε, διορθώνεται πλέον και ελπίζω έτσι να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Επιτροπής Εποπτείας της Όλαφ και αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα μπορεί να ασκεί καλύτερα η Επιτροπή Εποπτείας στα καθήκοντά της. Προκειμένου να πετύχουμε όμως όντω μία βελτίωση, πλέον θα πρέπει να μην ε, δημιουργηθούν άλλα προβλήματα ε, στην λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας. Θα πρέπει να εργάζεται, να συνεχίσει να εργάζεται η γραμματεία στους, ε, στα κτίρια της Όλαφ και να έχει πρόσβαση στα ε, έγγραφα και στα συστήματα IT. Και θα πρέπει επίσης ε, οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στη γραμματεία να προστατεύονται από σύγκρουση συμφερόντων και άλλα τέτοια μειονεκτήματα για την καριέρα τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει όλα αυτά να συμβούν πράγματα στην πράξη έτσι. Και δεν θα θέλω να σας πω ότι αυτή η μεταρρύθμιση ουσιαστικά αποτελεί και τεκμήριο ενός τεράστιου α, ε, λάθους. Αυτή η μεταρρύθμιση περιορίζει την παντοδυναμία του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ και είναι λυπηρό ότι αυτό ήταν απαραίτητο 17 χρόνια μετά τη σύσταση της ε, Όλαφ και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένδειξη έλλειψης επαγγελματισμού και έλλειψης ε, σωστής ε, διευθυντικής ικανότητας. Ε, πάντα υπήρχαν προβλήματα σε ό,τι αφορά την εποπτεία της Όλαφ, αλλά τόσο έντονα όσο ήταν αυτά τα τελευταίους 24 μήνες δεν ήταν ποτέ. Και έτσι λοιπόν αυτή η μεταρρύθμιση αποτελεί μία απάντηση και σας ευχαριστώ που όλοι συμβάλλετε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν με ακρίβεια το κατά πόσον η οδηγία της Όλαφ Όντως θα ενισχύσει τα δικαιώματα της Επιτροπής ε, ε, Εποπτείας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει άμεση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανεξάρτητα με τα, ε, τις ενστάσεις που αφορούν την ασυλία και τις ε, βελγικές έρευνες και θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα και με άλλα θέματα και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των ε, υπαλλήλων για να υπάρχει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και μεγαλύτερη ε, ε, ξε, μεγαλύτερος ξεκάθαρος χαρακτήρας σε ό,τι αφορά τις έρευνες της Όλαφ και για να λάβουμε υπόψη την εφιστάμενη κατάσταση. Αύριο λοιπόν σας παρακαλώ να υποστηρίξετε την πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λαϊκή Πρόεδρος. Και να δώσω τώρα το λόγο στην επιτροπή Γεωργέβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την εισηγήτρια, την κυρία Γκρέσλερ, για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να υποβάλει αυτή την πρόταση και αν τη συζητήσουμε σήμερα. Την υποβάλαμε στις 4 Μαρτίου, εμείς από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν μια πολύ ταχεία διαδικασία, κατ' εξαίρεση. Φτάσαμε στον κοινό μας στόχο τα τρία θεσμικά όργανα πολύ γρήγορα. Χθες ήμουνα στην Επιτροπή Εποπτείας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του καθώς και όλα τα μέλη για τη δράση που προωθήσαμε που στόχο έχει να εξασφαλίσει την εξαρτησία της Επιτροπής Εποπτείας διαχωρίζοντας τη γραμματεία της Επιτροπής και τον προϋπολογισμό από την ε, υπηρεσία που έχει λάβει την εντολή να εποπτεύει. Η Επιτροπή Εποπτείας ήταν πολύ δραστήρια, πρέπει να σας πω, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και τα μέλη άσκησαν τα καθήκοντά τους δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για την ανεξαρτησία της ε, Επιτροπής, μάλλον ότι η ανεξαρτησία της Επιτροπής ότι υποσκάπτεται. Αλλά υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και έχουμε ακούσει πολύ προσεκτικά και τους Ευρωβουλευτές και τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα βρούμε μια ξεκάθαρη λύση σε αυτό που θεωρείται πιθανός περιορισμό της ανεξαρτησίας. Και τι προτείνουμε λοιπόν για να το πω έτσι πολύ απλά και πρακτικά. Είναι ο προπολογισμό της Επιτροπής Εποπτείας ή μάλλον διορθώνει η ομιλήτρια. Έχουμε θέσει τον προπολογισμό της Επιτροπής Εποπτείας στα πλαίσια του PMO και τώρα και η γραμματεία εντάσσεται στο PMO από τη στιγμή που θα ισχύσει ο τροποποιητικός καονισμός. Ε, μιλάμε για μια προσαρμογή διοικητικής φύσεως, ούτως ώστε να διευκολύνουμε τις οργανωτικές και δημοσιονομικές πλευρές. Δεν θα επηρεάσουμε την ανεξάρτητη λειτουργία της Γραμματείας, ούτε της Επιτροπής, ούτε τον τρέχοντα προπολογισμό και το προσωπικό τους. Για να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά ξεκαθαρίζονται. Συμφωνήθηκε ότι η Κομισιόν θα κάνει μια δήλωση αύριο Είπα αυτή την έννοια και ελπίζω να ψηφίσετε επί της πρότασης. Εκφράζω την αποφασιστικότητα της Κομισιόν να κάνει ό,τι μπορεί για να ρυθμίσει τα θεσμικά θέματα που είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή μια επιτροπή εποπτείας θα πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της με ανεξαρτησία. Ευχαριστώ. Έχουμε υποβάλει λοιπόν, το PMO είναι η διοίκηση και η πληρωμή της Επιτροπής. Επίτροπε, Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα να ε, καλωσορίσω την ε, ε, λογική και το θάρρος, το κουράγιο της Επιτροπής να στηρίξει αυτό που φαίνεται λογικό, αλλά μετά από πιο προσεκτική εξέταση ε, φαίνεται σαν μια, ε, ένας περίεργος, ε, μια περίεργη μάχη που τελικά δεν θα έπρεπε να γίνεται αν όλα είχαν λειτουργήσει σωστά. Η Εποπτική Επιτροπή τη ΟΛΕΦ χρειάζεται μια ευρύθμη λειτουργούσα γραμματεία για να εκπληρώσει την αποστολή τη. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ανεξάρτητη από την ΟΛΕΦ η γραμματεία και η Εποπτική Επιτροπή. Άρα η χρηματοδότηση θα πρέπει να εξασφαλίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην εντάσσεται στον προπολογισμό τη ΟΛΕΦ. Αυτά είναι ε, ξεκάθαρα για μένα και χαίρομαι που συμφωνεί η Επιτροπή. Όμως, για αυτό το θέμα, αν η γραμματεία θα πρέπει να είναι παρούσα στο ίδιο κτίριο όπου με την Εποπτική Επιτροπή και με την Όλαφ, θα ήθελα να είμαι όσο το δυνατόν πιο ε, ξεκάθαρος γίνεται. Υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα στην Επιτροπή. Το να βγάλουμε τη γραμματεία από το κτίριο, χρησιμοποιώντας, προτάσσοντας σε μια τεχνητή επιχειρηματολογία, επιβεβαιώνει την κατάσταση στην Όλαφ. Η Όλαφ πρέπει να ασχολείται με την έρευνα υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης. Δεν θα πρέπει να ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Η Αποτελεσματική Επιτροπή της Επιτροπής ε, προϋποθέτει ότι θα υπάρχει διαρκής επαφή με την Όλαφ η γραμματεία θα πρέπει να παραμείνει στο κτίριο της Όλαφ. Συγχαρητήρια προς την ε, εισηγήτρια, διότι φρόντισε να επικρατήσει η κοινή λογική. Σας ευχαριστούμε. Αγιάλα Σέντερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ταχύτατη τροποποίηση του κειμένου, του κανονισμού που θέλει να ρυθμίσει ένα πρόβλημα πολύ πιο ευρύ και περίπλοκο ε, και που έχει να κάνει με τις σχέσεις ανάμεσα στην Όλαφ και την Επιτροπή Εποπτείας. Ε, αυτή η περίπλοκη σχέση ε, υπάρχει εδώ και χρόνια γιατί έχουμε διαπλοκές επαγγελματικέ, προσωπικές και δημιουργούμε μια πολύ βαριά κατάσταση. Δημιουργήθηκαν ακόμα και προβλήματα και καυγάδες μέχρι που ε, αφαιρέσαμε την ασυλία του διευθυντή της Όλαφ. Μέχρι αυτού του σημείου φτάσαμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι, ότι αυτή τη στιγμή ανακτηθεί αυτή η ανεξαρτησία, η Επιτροπή Εποπτείας θα μπορέσει να ξανακάνει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της Όλαφ σε σχέση με την Επιτροπή και σε σχέση με οποιαδήποτε άλλα θεσμικά όργανα. Να σεβαστεί την προστασία των δεδομένων με απόλυτη αυστηρότητα, τελευταίως είχαμε αμφιβολίες, καθώς και να ε, εξασφαλίσει τα δικαιώματα, τα δικονομικά δικαιώματα των ανθρώπων που βρίσκονται υπό έρευνα από την Όλαφ. Η ταχύτητα αυτή ήταν πάρα πολύ θετικό πράγμα, αλλά πρέπει να λύσουμε όλα αυτά τα σύνθετα προβλήματα και θα πρέπει να δώσουμε στη γραμματεία της ε, Επιτροπής Εποπτείας ένα νέο στάτους, μια ανεξαρτησία που θα ήθελα να σας ρωτήσω κυρία Αντιπρόεδρε, με ποιο τρόπο τα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας θα λογοδοτούν. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι πραγματικά αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιον λογοδοτούν. Ε, σε, μέσα σε ποιο πλαίσιο αυτή τη στιγμή, σε ε, ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες. Ο κύριος Άρνοτ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ασφαλώς είναι πολύ βασικό ε, η υπηρεσία κατά της απάτης να είναι αμερόληπτη. Αυτό προφανώς ε, θα συμβάλλει στην αξιοπιστία της ε, και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Και η γραμματεία της θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Και για μία φορά θα πρέπει να σας πω ότι οι τροπολογίες της Επιτροπής φαίνεται να έχουν ε, τη σωστή πρόθεση. Να είναι απόλυτα σαφές το ότι θα πρέπει να πετύχουμε την ανεξαρτησία και ότι θα υπάρχει παρέμβαση της Επιτροπής στην ε, διαδικασία εποπτείας της Επιτροπής Εποπτείας. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία. Το κατά πόσον αυτό πάει αρκετά μακριά και κατά πόσο είναι αρκετά ξεκάθαρο και διαυγές το θέμα της μη παρέμβασης και της ανεξαρτησίας, αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λεμπρετών για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, την Όλαφ την δημιούργησαν μετά την πτώση της Επιτροπής ε, πριν από 17 χρόνια. Ε, θα λειτουργούσε ως το ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής σε πλήρης αποτυχία, διότι παραβιάζεται το εκμήριο της αθωότητας προσφάτως η διπλωματική ασυλία του Διευθυντή ε, ακυρώθηκε μετά από την αίτημα των βελγικών αρχών. Προς το παρόν δεν μπόρεσε να ασκήσει η υποπτική αρχή της Όλαφ για δύο λόγους. Ο πρώτον γιατί εξαρτάται από την Όλαφ και διαχειρίζεται η Όλαφ τον προϋπολογισμό και ε, ε, επίσης δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα. Είναι σκάνδαλο. Χαίρομαι λοιπόν διότι με το σημερινό έγγραφο που προτείνεται να αναβαθμιστεί ο ρόλος της υποπτικής Επιτροπής ε, πολλαπλασιάζονται όμως ε, οι καταχρήσει εξουσίας από πλευρά της Όλαφ, πώς πρέπει να την καταργήσουμε και να ξεκινήσουμε πάλι πάνω σε μια υγιή βάση δημιουργώντας ένα νέο οργανισμό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόρβιν Μίκεν. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος ε, έκανε μάλλον ε, ένα αστείο, διότι πριν από ένα χρόνο είπαμε ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή εισαγγελία και ότι η Όλαφ δεν μπορεί να κάνει δικές της έρευνες. Βλέπουμε όμως πως οι καταχρήσεις εξουσίας γίνονται από την Όλαφ, η άρση της ασυλίας του διευθυντή που δεν είναι σίγουρη, ε, το αποδεικνύει αυτό και έχουμε ε, κατηγορίες από πλευράς ε, τριών επιτροπών και τώρα Μας λέτε ότι το Μάρτιο ξεκίνησε η διαδικασία αναθεώρησης και τώρα ε, από όλα αυτά το πρόβλημά μας είναι αν θα είναι η γραμματεία στο ίδιο κτίριο ή όχι. Όχι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι αντικατάσταση στις εποπτικές αρχές, ριζοσπαστική δράση και όχι το που θα να μας απασχολεί, που θα είναι η γραμματεία. Ο κύριος Σεντόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που έχω ήδη πει και θα ήθελα να επαναλάβω και αυτά που είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πριν από εμένα. Αλλά αγαπητέ κυρία Επιτροπέ, θα ήθελα να τονίσω το εξή. Η διαφάνεια και η ακαιρεότητα αποτελούν κοινέ μας προτεραιότητες. Αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο και όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητοι υπηρεσίες, ανεξάρτητες υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπεράνω κάθε υποψίας ε, και με απόλυτη ανεξαρτησία θα μπορούν να ερευνούν περιπτώσεις απάτη. Ε. Και αυτό ισχύει λοιπόν ε, για τους κόλπους της ΟΛΑΦ, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, καθώς και η Επιτροπή Εποπτείας, προκειμένου να μπορέσει να παρέμβει σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά στους κόλπους της ΟΛΑΦ. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή Εποπτείας ε, και η γραμματεία είναι ουσιώδου σημασίας και αυτές λοιπόν οι δύο υπηρεσίες θα πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητες από την όλα για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ και καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πιτέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία για την εποπτική αρχή της ΟΛΑΦ. Προς το παρόν ε, έχουμε αμφιβολίες σε σχέση κυρίως με το θέμα της σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Ε, όταν ε, το προσωπικό και η χρηματοδότηση μιας εποπτικής αρχής συνδέεται με τον οργανισμό που πρέπει να εποπτεύει είναι φυσικό αυτό και ε, γι' αυτό θα πρέπει να εκπληρωθούν αυτές, αυτά τα αιτήματα που έχουν εκφραστεί για τη μεγαλύτερη ανεξαρτησία της εποπτικής αρχής διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται αντικειμενικά η εποπτεία της Όλαφ. Ε, η μεταφορά τώρα της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κατοχυρώσει την ανεξαρτησία της εποπτικής αρχής και ευχαριστούμε την Επίτροπο Γεωργίευα που εισάκουσε τις αιτήσει του Κοινοβουλίου. Η διαδικασία κάτι θεά υπόσπιση. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να σας πω ότι ακούσαμε μεγάλη προσοχή τη συζήτηση αυτή στην τσεχική δημοκρατία. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τέτοια ζητήματα ανεξαρτησίας. Δεν είναι θεωρητικό το ζήτημα αυτό για μας. Για παράδειγμα, ε, τέθηκε το θέμα της ε, Πρωθυπουργού και δεν επιλύθηκε. Και οι συγκρούσεις αυτές ακριβώς την όλα αυτή λευκάνθηκαν. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα πρέπει η πρεσία αυτή να είναι ανεξάρτητη προκειμένου και η τσεχική κοινή γνώμη να μπορέσει να αποδεχτεί και τις αποφάσεις σε ό,τι αφορά την ε, Πρωθυπουργό Τίθεται λοιπόν θέμα πολιτικής ε, σταθερότητας ε, για την τσεχική δημοκρατία. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια, ευχαριστώ και την Επίτροπο για το γεγονός ότι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό. Εξ των ε, εκλογέων μας πρέπει να σας πω ότι δεν πρόκειται για ένα θερτικό πρόβλημα αυτό το θέμα της ανεξαρτησίας. Έχει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές συνέπειες για μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαγιάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Όλαφ είναι κρίσιμη υπηρεσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια. Έτσι η Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ καθώς και η γραμματεία της πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν αυξημένη ανεξαρτησία προκειμένου να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση συμφερόντων ταυτόχρονα η όλαφ ως ειδική ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης θα πρέπει να συνδυάσει τη διαφάνεια με την αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής άλλωστε το σύνολο των παρατυπιών που αναφέρθηκαν για το 2014 ανέρχεται περίπου σε τρία δισεκατομμύρια ευρώ ενώ ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των παρατυπιών που δηλώθηκαν είναι κατά 36% έξι μεγαλύτερος σε σχέση με το 2013, χιλιάδες γεγονός που δείχνει ότι η όλαφ δεν έχει κάνει τίποτα για να συμβάλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών εταιριών. επομένως εκτός από την ανεξαρτησία της επιτροπής εποπτείας και της γραμματείας της αυτό που προέχει είναι η όλαφ να αποκτήσει ένα πιο ενεργό ρόλο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών καθώς και κάθε παράνομης δραστηριότητας που λαμβάνει η χώρα στην ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Επίτροπος Γεωργίευα έχει το λόγο. Thank you very much. Uh, ευχαριστώ για τα σχόλια που εκφράσατε. Ακούστηκαν ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς για τη γραμματεία. Για το αν θα συνεχίσει να εδρεύει στο κτίριο της Όλαφ. Σα επιβεβαιώνω πως ναι, η γραμματεία όντω θα συνεχίσει να εδρεύει στα κτίρια της ΟΛΑΦ και θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση στις πληροφορίες από πλευράς της. Εκφράστηκε μια ανησυχία επίσης ότι η γραμματεία θα ενσωματωθεί στην Επιτροπή. Το θέμα των πόρων το έχουμε εξετάσει σοβαρά. Έχουμε δει διάφορες δυνατότητε. Έχουμε δει τις υπηρεσίες ανθρωπίνων πόρων μας. Έχουμε δει την ε, Γενική Γραμματεία, έχουμε δει, δει το PMO και τελικά επιλέξαμε το γραφείο ε, των υπηρεσιών πληρωμής γιατί δεν έχουν καμία ευθύνη περί πολιτικής. Και εκεί μπορεί να δώσουν μπορεί να ε, δώσουν άσυλο στη γραμματεία. Μπορεί να υποδεχτούν αυτή τη γραμματεία. και μπορούν οι άνθρωποι εκεί να έχουν τα γραφεία τους χωρίς να υπάρχει καμία ανάμειξη στη δουλειά τους. Ο επικεφαλής της ε, γραμματείας ασχολείται με το θέμα αυτό. Κοιτάξαμε όλες τις υπηρεσίες και θεωρήσαμε ότι είναι το πιο ουδέτερο πόστο. Εκεί δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Είναι το καλύτερο μέρος που μπορούμε να βρούμε. Γι' αυτό αποφασίσαμε να το επιλέξουμε. Επίσης, Ακούστε ένα σχόλιο ότι είναι σημαντικό το που εδρεύει η γραμματεία, αλλά ακόμα πιο σημαντικό όμω είναι η σύνθεση τη επιτροπή ε, Εποπτεία. Και ορισμένοι είπαν ότι πρέπει να υπάρξουν αντικαταστάσει στην Επιτροπή Εποπτείας. Κυρία Γκρέστερ, ξέρει πολύ καλά ότι προσπαθήσαμε να δούμε ποια θα είναι τα μελλοντικά μέλη της Επιτροπής Εποπτείας και ψάξαμε να βρούμε τα κατάλληλα άτομα από τα τρία θεσμικά όργανα Πρόσφατα συμφωνήσαμε πάνω σε πέντε νέα μέλη που θα αναλάβουν τις αρμοδιότητές τους τη στιγμή που θα εκπνεύσει η θητεία των σημερινών μελών. Έχουμε επίσης και μία ε, λίστα με επιπλέον 7 άτομα που είναι πάρα πολύ ικανά και νομίζω ότι θεσμικά είμαστε σε πολύ καλή θέση. Μπορούμε να φτιάξουμε μία επιτροπή εποπτείας πολύ ικανή για να κάνει τη δουλειά που της έχει επιφορτιστεί. Για το πώς θα λάβει χώρα η μετάβαση. Δεν το έχουμε σκεφτεί πολύ, γιατί πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που θα πάρουν αυτές τις θέσεις και θα μπουν σε αυτή τη λίστα των πέντε ατόμων, καθώς και στην λίστα των απληρωματικών μελών, των 7 δηλαδή, είναι απόλυτα ικανά μέλη και τις επόμενες μέρες η διαδικασία επιλογής θα οριστικοποιηθεί. Θα επιλέξουμε τους, τα άτομα αυτά με καλή συνεργασία ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα. Ευχαριστούμε την Επίτροπο και τώρα η, Επίτρο, η συγγήτρια, συγγνώμη, η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που έκαναν παρατηρήσεις Όλοι έχετε λίγο δίκιο, γιατί όντως πρόκειται για ένα πολύ περιπλοκό θέμα. Και κυρία Αντιπρόεδρε, είσαστε η πρώτη επίτροπο που πραγματικά επέλυσε ένα πρόβλημα. Ή τουλάχιστον που προσπάθησε να το επιλύσει. Προσπαθήσαμε κι εμεί να το επιλύσουμε, αλλά α μην ξεχνάμε ότι σήμερα πρόκειται για μια νέα σημαντική αφετηρία σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Εποπτεία. Και αυτή η νέα ε, κίνηση ελπίζουμε ότι θα κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι θα δώσει τις σωστές ε, λύσεις. Και εδώ θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά που είπε και η συνάδελφη, η συνάδελφος Αγιάλα. Σε ποιον λογοδοτεί η Επιτροπή Εποπτείας σε εμάς ε, και εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να φροντίσουμε ότι κάνει σωστά τη δουλειά της και γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν μια καλή σχέση αξιόπιστη σχέση με το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Δεν ε, μπορούμε να αφαιθούμε σε φιλοσοφικές σκέψεις. Θα πρέπει να συνεχίσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να θελεχώσουμε σωστά την εταιρεία και πώς μπορούμε να καλύψουμε τα κενά τα νομικά. Και σε αυτά συγκαταλέγεται και η πρόσβαση της Επιτροπής στα έγγραφα θα πρέπει να λαμβάνουν και τις εκθέσεις της Όλαφ γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κατηγορίες τις οποίες να μην γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι. Νομίζω λοιπόν ότι πλέον έχουμε κάποιες σημαντικές εμπειρίες τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη μεταρρύθμιση της Όλαφ σε ό,τι αφορά την εισαγγελία, σε ό,τι αφορά μια νέα θεσμική διαμόρφωση της όλα αυτή συνεργασία με έναν ευρωπαϊκό, ευρωπαίο εισαγγελέα. Ξέρουμε λοιπόν προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε για να πετύχουμε μια πραγματική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Γκρέσλα και έτσι όλο